Μετά τα ε, διαδικαστικά, μετά τις ανακοινώσεις. Όπως γνωρίζουμε, ο κύριος Σταύρος Λαμπρινίδης μου διεβίβασε τη συμμετοχή του στην ελληνική κυβέρνηση από τις 17 ε, Ιουνίου 2011. Το Κοινοβούλιο σημειώνει την ανακοίνωση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ε, κανονισμού για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα υπόλοιπα αντίστοιχα ε, άρθρα διαπιστώνει τη χειρία από τις 17 Ιουνίου 2011. We will continue uh, with our work συνεχίζουμε και ευχόμαστε τον πρώην συνάδελφο καλή τύχη και ό,τι καλύτερο. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Δημητρίου Βρούτσα που θα δικαστήσει τον κύριο Λαμπρινίδη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το διαπιστώνει το Κοινοβούλιο και ε, τίθεται σε ισχύ αυτή ε, ε στις 22 Ιουνίου 2011. Καλώς όρισε ο καινούριο συνάδελφος. Και μέχρι την έγκριση ε, της εντολής και των διαπιστευτήρων ε, θα πρέπει να υπογράψει και ε, τη δήλωση ότι δεν υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου. Και μέχρι τότε ο κύριος Ρούτσας θα ε, συνεδριάζει στο Κοινοβούλιο εξ όλα τα όργανα και θα απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τη θέση του Ευρωβουλευτού. Και καλή τύχη ευχόμαστε επίσης και στο νέο συνάδελφο. Μα ακούτε, διαδικαστικό. Δεν θυμάμαι το άρθρο γιατί δεν έχω τον κανονισμό μαζί μου. Αλλά βλέπω ότι έχουν πολιτικές αφήσει στην άλλη πλευρά του ημικυκλίου. Αυτό είναι κατά του κανονισμού. Δεν με πειράζει εμένα προσωπικά, αλλά επανειλημμένα έχω ζητήσει στο Κοινοβούλιο και βλέπω ε, ότι δεν ε, ισχύει να ε, έχουμε ίση μεταχείριση προς όλους. Εάν αφήνετε αυτές τις αφήσει, εγώ θέλω να βάλω την αφήσα του UKIP. Μπορούμε να αποφασίσουμε κάποια στιγμή προς τη μία κατεύθυνση την άλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάτεν που με έφυσα την προσοχή τόσο σαφώς για τις αφήσει παρακαλώ ε, να τις αφαιρέσετε συνάδελφοι από τα έδρανά σας. Παρακαλώ απομακρύνετε τις αφήσει αυτές. Σας παρακαλώ. And then we can continue with our work. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Κυρία Λίν. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τους διαδηλωτές, νομίζω ότι είναι τελείως λάθος να επιτρέπεται να μπαίνουν στο κοινοβούλιο και να εμποδίζουν τους βουλευτές να μπουν να ψηφίσουν. Ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος και του αιτήματο. κάτι πρέπει να γίνει να βεβαιωθούμε ότι οι βουλευτές θα μπορούν να μπαίνουν να ψηφίζουν χωρίς να τους εμποδίζει κανείς. Ευχαριστώ κυρία Λίν. Θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Μάτλενε. ναι, ευχαριστώ πρόεδρε πολύ. Θα ήθελα να σας αναφέρω μια χαρμόσυνη είδηση. Ο Χέρτ Βίλντερ σήμερα το πρωί ε, εθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες ο ηγέτης του κόμματός μου ε, που τον βάρεναν ε, η ελευθερία του λόγου στην Ολλανδία διαφυλάσσεται πρόεδρος Διακόπτη. Τι σχέση έχει αυτό με τις εργασίες μας εδώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές ψηφοφορίες. έχουμε και γραπτή δήλωση πρώτα απ' όλα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE